Good morning everybody. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίασή μας. is always Το πρώτο θέμα όπως πάντα η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Και τώρα η ανακοινώσει του Προέδρου. Έχουμε τον ορισμό των εισηγητών. Η κυρία Ανθία Μακιντάιρ έχει οριστεί η συγκήτρια για την πρόταση οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων κατά των απατών που αντικαθιστά την απόφαση πλαίσιο του Συμβουλίου 2000 383 κάθετος τσα. Ο δε κύριος Τιμόθεος Κίρκοφ έχει οριστεί εισηγητής για μια πρόταση κανονισμού για διάφορα θέματα πλήρωμα. Ο δε κύριος Κλέης έχει οριστεί εισηγητής επίσης για το θέμα των οργανώσεων με τις οποίες έχει συνάψει συμφωνίες η Ένωση, κυρία Μπένοβα, η για την έκθεση της ΝΟΜ η Γιούρη για τον έλεγχο από τα κράτη-μέλη κλπ. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, δεν ακουστούν αντιρρήσει μέχρι το τέλος της συνεδρία, τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Δηλαδή, 3 Σεπτεμβρίου 2012, 8 Δεκεμβρίου 2011, 29 Νοεμβρίου 2011, 31 Αυγούστου 2011, 20 Απριλίου 2011 και 28 με 29 Σεπτεμβρίου 2010. Αυτά ήταν οι ανακοινώσει. Και τώρα θα αρχίσουμε την κανονική μας εργασία με κοινή συζήτηση. Έχουμε το θέμα της απαλλαγής 11. Σε πολλά θέματα θα σας τα διαβάσω. Γενικό προϋπολογισμός τμήμα 3 Επιτροπή. Ευρωπόλ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για τη Διαχείριση της Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα Frontex, το ΣΕΠΟΛ, η Ευρωδίκ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιτήρησης Ναρκωτικών, η Υπηρεσία για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, ο Γενικός Προϋπολογισμός για την Προστασία των Δεδομένων, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος και για όλα αυτά, για όλες αυτές τις γνωμοδοτήσεις, συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Γεώργιος Παπα-Νικολάου του ΕΛΚ. Βέβαια έχουν κατατεθεί και τροπολογίες. για τις γνωμοδοτήσεις αυτές του κυρίου Παπα-Νικολάου και πρώτα θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για τις αρχικές του δηλώσεις και μετά θα γίνει η ανταλλαγή των απόψεων. Την περασμένη εβδομάδα έληξε η διορία κατάθεση τροπολογιών. Δεν έχουν ακόμα γίνει όλες οι μεταφράσεις, αλλά θα γίνουν. Κύριε Παπα-Νικολάου μου, λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από δύο εβδομάδες είχαμε την αρχική εισαγωγή των ε, σχεδίων γνωμοδοτήσεων για τα ζητήματα αυτά. Μετά συζητήσαμε τις τροπολογίες και όντως δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να γίνουν οι μεταφράσεις, όμως εάν όποιο, όποιος συνάδελφος θέλει διευκρινήσεις είμαστε στη διάθεσή του να εξηγήσω. Καταρχάς, να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες, την κυρία Μακοβέ, την κυρία Κόνσια, για Κολίνο, για τους υπόλοιπους συναδέλφους. Δεν έχουμε πολλές τροπολογίες για όλες τις εκθέσεις, τις γνωμοδοτήσεις. Εννέα γνωμοδοτήσεις και περίπου 60 τροπολογίες. Και από ό,τι μαθαίνω κάποιες θα αποσυρθούν κιόλα. Για κάθε γνωμοδότηση έχουμε ορισμένες τροπολογίες, αλλά ενδέχεται να γίνουν αλλαγές σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες. Θα αναφερθώ σύντομα σε κάθε γνωμοδότηση ακολουθώντας την ημερήσια διάταξη. Ωστόσο, πριν θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένες τροπολογίες που υπέβαλε ο ίδιος για να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Τον έλεγχο των ευρωπαϊκών οργανισμών. Πριν από δύο εβδομάδες, όταν πρωτοσυζητήσαμε στο ελεκτι... εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου, προ... Ε, ύψιστη προτεραιότητα ήταν να προσπιστούν τα συμφέροντα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και μου ζητήθηκαν διευκρινήσεις, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, να πω ότι η παράγραφος αυτή απευθύνεται στο ελεκτικό συνέδριο. Δηλαδή, περιμένουμε περισσότερα από το ελεκτικό συνέδριο, περισσότερη δουλειά και όχι από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Εμείς ως Κοινοβούλιο χρειάζεται να έχουμε όσο δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και ως Επιτροπή, όπως αναφέρε και η Πρόεδρος, οι απαλλαγές για τις ε, προναφερθήσεις υπηρεσίες, για τη Frontex, για τη Europol, τη Cepol, τη Eurojust, οργανισμός ε, για τα θεμελιώδη δικαιώματα, ναρκωτικά. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο για σχόλια. Να πω όμως ότι αρκετές ε, τροπολογίες θα αρχίσω μάλλον με την πρώτη γνωμοδότηση. Υπάρχει πρόταση διαγραφής της παραγράφου 3 για την πολιτική για τις θεωρήσεις και την ελεύθερη ε, μετακίνηση των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την Europol, υπάρχουν ορισμένε τροπολογίες που αλλάζουν το ύφος της γνωμοδότησης. Συμφωνώ με την ε, συνάδελφο κυρία Ματιέ για το θέμα αυτό. Η Europol έχει κάποια προβλήματα όπως ανέφερε το ηλεκτρικό συνέδριο και αυτό όμως ε, είναι φυσιολογικό, είναι στα όρια του φυσιολογικού διότι η Europol είναι μια νέα υπηρεσία. Ωστόσο θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας της. Η Europol έχει αναλάβει πολλά και διαφορετικά έργα και ο φόρτος κατέστησε δύσκολο στην Europol να τα απεξέλθει πλήρω σε, όλες, σε όλα αυτά που είχε να κάνει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το ΕΛΚ για τη συνεργασία τους και να ευχαριστήσω και όλους για τις επιστολές τους καθώς και τον διευθυντή της Europol. Νομίζω η τροπολογία 5 ε, είχε ένα πρόβλημα. Έχουμε βρει όμως μία λύση και δεν θα πρέπει να υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες. Τώρα, για την γνωμοδότηση Frontex, πιστεύω ότι η τροπολογία 3 της κυρίας Κέλλερ ανταποκρίνεται στο σκεπτικό της τελευταίας πρότασης της παραγράφου 2. ΣΥΠΟΛ. Πολύ σημαντική είναι η τροπολογία 9 πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ΣΥΠΟΛ θα συνεχίσει να εργάζεται στα γραφεία της μέχρι το Μάρτιο του 2013. Ωστόσο, πρέπει να διασφαλιστεί ομαλή συνέχεια και μετά την ημερομηνία αυτή. Προτείνω να διαγραφεί η τροπολογία, με την τροπολογία 11 η παράγραφος 4. Επίσης υπέβαλα γλωσσική, τροπολογία γλωσσικού ύφου στην παριθμόν 12. Τώρα, όσον αφορά το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, οι περισσότερες τροπολογίες αναφέρονται στις εργασίες της υπηρεσίας αυτής. Επίσης, η κυρία Μακοβέη με ενημέρωσε ότι θα αποσύρει ορισμένε τροπολογίες της στη γνωμοδότηση αυτή. Τώρα, όσον αφορά τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουμε τις τροπολογίες 5 και 6 που αφορούν περιπτώσεις παρενόχλησης η κυρία Ματιέ και η κυρία Μακοβέη ενημέρωσαν τη γραμματεία σχετικά. Είχαμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό και σύμφωνα με τις νέες πληροφορίες θα γίνει προφορική τροπολογία στις τροπολογίες που έχουν ήδη υποβληθεί γραπτός. Επίσης ε, στις τροπολογίες που αφορούν την εποχή εικόν. Και τέλος, η γενική γνωμοδότηση για όλες τις οι υπηρεσίε από την ε, η κυρία Γκόντ και η κυρία Ματιέ ανέφεραν τις πιθανές συγχωνεύσεις οργανισμών και το γεγονός αυτό ενδεχομένως επηρεάσει αρνητικά το έργο τους. Συζητήσαμε με την Επίτροπο κυρία Μάλιμστρομ και στη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο της Επιτροπής μας κύριο Αγγιλάρ για την σημασία που έχει το θέμα. Επίσης, να χαιρετήσω την τροπολογία 4 της κυρίας Κέλλερ. Τέλος, να ολοκληρώσω ευχαριστώντας θερμότατα κάθε έναν από εσά και κάθε οργανισμό για την συνεργασία και τις συνεισφορές σας στο σχέδιο αυτό Θα χαρώ πολύ να συνεργαστώ με όλους τους ενδιαφερομένους και με όλους τους συναδέλφους έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια οριστική μορφή της έκθεσης. Να ευχαριστήσω και την Γραμματεία και την κυρία Χιούμπερ και όλους σας για τα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Παπα-Νικολάου. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Λίγες παρατηρήσεις έχω να κάνω και ερωτήσεις. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες που, αφοράν, που αφορούν συγγνώμη, την ε, συγχώνευση Europol και Eurosea. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να περάσει στη γενική απαλλαγή για τον προϋπολογισμό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ε, να το συζητήσει κανείς αυτό το θέμα στα πλαίσια το δημοσιονομικά γιατί δεν είναι ένα απλά οικονομικό θέμα, είναι πολιτικό. Κάτι που μοιάζει με το προηγούμενο αφορά την υπηρεσία για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Διαρωτώ με αν η διαδικασία απαλλαγή είναι ο καλύτερος τρόπος να το αντιμετωπίσουμε ή αν έχουμε κάποιον άλλο τρόπο, δεν ξέρω ποιον. αλλά μια απαλλαγή τη δίνει κανείς ή δεν τη δίνει. Οπότε αν αρχίσουμε να το συζητάμε αυτό το θέμα στα πλαίσια της απαλλαγής, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αποκλειστικά τον προϋπολογισμό. Φυσικά έχει σχέση, αλλά δεν είναι αποκλειστικά δημοσιονομικό. το ότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις υπηρεσίες αυτές ε, να ξεπερνούν, αν θέλετε, τον ετήσιο δημοσιονομικό χαρακτήρα τους. Προβλέπετε μερικές φορές να μην χρειάζεται ένας διαθωτικός προϋπολογισμός, Οπότε στην περίπτωση του διορθωτικού προϋπολογισμού ο ρόλος της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι φυσικά πολύ πιο περιορισμένος από ότι στα πλαίσια του κανονικού περιορισμού εμένουμε στην αρχή του ετήσιου χαρακτήρα των προϋπολογισμών. Το συζητάμε αυτό σε μόνιμη βάση. Κάθε χρόνο ξαναρχόμαστε στην ίδια συζήτηση. Σε μία υπηρεσία βλέπουμε να έχει σημειωθεί πρόοδο σε σχέση με την ανάκτηση του ετήσιου χαρακτήρα, ενώ άλλες πάλι μας πηγαίνουν πίσω. Είναι ένα πρόβλημα γενικότερο χαρακτήρα όταν βλέπουμε η Επιτροπή να χρηματοδοτεί θέματα πάνω στα οποία δεν έχουμε εκφραστεί. Εμείς είχαμε πει ότι δεν θα έπρεπε σαν παράδειγμα να υπάρξει χρηματοδότηση ορισμένων ταμείων. Θα μπορούσαμε, είχαμε πει εμείς, να κάνουμε κάποιες προβλέψεις ε, για επιμέρους δημοσιονομικές ρυθμίσεις, αλλά η Επιτροπή μας είχε κατά κάποιο τρόπο αγνοήσει και δεν ξέρουμε πού ακριβώς έχουμε καταλήξει σε τέτοια θέματα. Ευχαριστώ κύριε Γκέπχαρτ. Κύριε Άιντφελτ. Καταρχήν για την υπηρεσία θεμελιωδών. Διαφωνώ και με την κυρία Κέλλερ ότι δεν είναι εδώ το κατάλληλο πλαίσιο για να τεθεί το θέμα των παρενοχλήσεων ή των ερευνών της Όλαφ η υπηρεσία των θεμελιωδών πρέπει να τα διασαφηνίσει όλα αυτά. Το θέμα συζητιέται πολλά χρόνια. Και αν, όπως λέει ο διευθυντής της, όλα πάνε καλά, τότε να έρθει να μας το εξηγήσει. Μια για πάντα. Δεύτερον για την Ευρωπόλ. Ο συντάκτης, ο εισηγητής είπε ότι είναι καινούριο θεσμός και άρα έχει ορισμένα θέματα προϋπολογισμού που είναι θεμητό να υπάρχουν αλλά δεν είναι και τόσο καινούργιο ο τελικά. Και τέλος το τελευταίο που είπε η κυρία Κέλλερ για την τάση που σημειώνεται να συμπεριλαμβάνονται στον προϋπολογισμό χρήματα για θέματα που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί αποφασιστεί. Γι' αυτό δεν φταίνουν οι υπηρεσίες αλλά η Κομισιόν που έδωσε 50 εκατομμύρια ευρώ για εθνικά προγράμματα στοιχείων επιβατών πράγμα το οποίο μπορεί τεχνικά να είναι σωστό αλλά ηθικά απαράδεκτο. Η κυρία Κέλλερ θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, να εξηγήσω στη Σοφή, συμφωνώ για, τα θεμελιο... για την υπηρεσία θεμελιωδών, αλλά εγώ ήθελα να ερευνήσω αν δεν θα έπρεπε να έχουμε αποσαφηνίσει από τους διευθυντές και από άλλες υπηρεσίες άμα είναι σωστά αυτά που είπες. Κύρκο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τα σχόλια που ήθελα να κάνω αφορούσαν τις συγχωνεύσεις υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων αυτών. Μερικές από αυτές τις υπηρεσίες δεν μας έδωσαν απολογισμό και αποτελέσματα σαν και αυτά που θα επιθυμούσαμε και αυτό το δείχνει και το ελεκτικό συνέδριο, η Ευρωπόλα, ας πούμε την οποία έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία είναι πολύ σημαντική υπηρεσία, αλλά έχουν ακουστεί επικρίσεις. Και για τον απολογισμό και τη διαχείρισή της. Επομένως, δέχομαι με την εργασία του εισηγητή, αλλά πρέπει να το ξαναδούμε λίγο ακριβέστερα. Τώρα το κατά πόσον το ελεγκτικό συνέδριο καθόρισε κριτήρια που οδηγούν στις επικρίσεις όπως λέμε γενικά για τις απαλλαγές ποιες είναι αυτές οι επικρίσεις είναι σημαντικές ή απλώς τεχνικές λεπτομέρειες θα με διέφερε ιδιαίτερα λοιπόν να τα μάθω αυτά γιατί διστάζω να δεχτώ επικρίσεις της Ευρωπόλ που δίνουν την εντύπωση ότι είναι, υπάρχουν σημαντικές δυσλειτουργίες. Νομίζω ότι το ελεγκτικό συνέδριο θέτει τεχνικά καθαρά κριτήρια και φραγμούς. Να μην υπερβάλλουμε λοιπόν, αλλά ας τα δούμε να ξέρουμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκοπ. Η γραμματεία μου είπε μόλις ότι προβλέπεται να έρθει ο διευθυντής της υπηρεσίας θεμελιωδών για να μας τα αποσαφηνίσει αυτά. Η Κομισιόν μήπως τώρα θα ήθελε να μας πει τίποτα. Αν όχι. Α, ναι για την απαλλαγή της Κομισιόν. Κατατέθηκε μία τροπολογία της κυρίας Κίνγκα Γκέντς. Δεν έχουμε σχόλια. Σημειώνουμε το αίτημα της Επιτροπής σας να βελτιώσουμε τον δημοσιονομικό μας σχεδιασμό. Για το 11 πάντως οι αριθμοί είναι αυτή που είναι και για το 12 φαίνεται ότι υπάρχει πολύ μεγάλος ρυθμός απαρόφησης. Ο εισηγητής. Να διευκρινίσω αυτό που είπα για την Europol και να απευθυνθώ στην κυρία Ιντφέλντ. Η Europol είναι ένας καινούριος οργανισμός. Αυτό εννοούσα και ίσως παρεξηγήθηκα και ως ένας νέος οργανισμός που λειτουργεί από τον Ιανουάριο ε, του 2010. Είναι ένα οργανισμό και αυτό το επιχείρημα χρησιμοποιεί και η ίδια η Europol για να δικαιολογήσει. Κύριε Κέλλερ, ε, ξέρω πως δεν είναι εύκολο να διεξάγουμε πολιτική συζήτηση στα πλαίσια των απαλλαγών και δεν έχουμε όντως περιθώρια ευελιξίας για τροπολογίες και για πολιτικές συζητήσεις όταν αυτό είναι κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο, που πρέπει να το κάνουμε και να εστιάσουμε αυστηρότατα στον προϋπολογισμό των οργανισμών αυτών. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με αρμόδιους και να βρούμε κάποια ισορροπία και το αναλύσαμε αρκετά. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι κατά τη διάρκεια της κατάρτισης της γνωμοδότησης αυτής συνειδητοποίησα ότι όταν ένα θέμα προκύπτει στην Επιτροπή μας και ενημερωνόμαστε και οι συνάδελφοι υποβάλλουν τροπολογίες, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε τα θέματα αυτά, ιδιαίτερα όταν η έκθεση αυτή είναι η αφορμή για συζητήσεις για μετά την απαλλαγή. Όντως όμως κάποια σχόλια Πολύ σωστά είπατε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότηση. Έτσι ώστε να έχουμε και ένα μπούσουλα για το μέλλον και τις ε, συζητήσεις που θα κάνουμε. Προσπαθούμε λοιπόν να επιτύχουμε μια ισορροπία χωρίς να ξεχνάμε και τη δουλειά που κάνουμε εδώ. Την κατάρτιση δηλαδή γνωμοδοτήσεων για τον και απαλλαγών για τον προϋπολογισμό. Και θέλω πραγματικά να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο προϋπολογισμό και μόνο. Και αυτό προσπάθησα να κάνω εδώ. Τώρα, η συγχώνευση Europol και Σίπολ. Συμφωνώ πως αυτό το θέμα δεν είναι κάτι που απαραίτητα πρέπει να θίξουμε στις ε, εκθέσεις απαλλαγή. Όμως, όταν συζητείτε το θέμα, όταν έχουμε τροπολογίε. Πρωτοβουλίε, επικοινωνία με τις επιτροπές, ανακοινώσει και από την Κομισιόν, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι πολιτικά μας απασχολεί αυτό το θέμα. Αυτό προσπαθήσαμε και όλας να διαφανεί στο κείμενο. Συμφωνώ ότι είναι ένα θέμα που δεν θα τελειώσει εδώ και θα το συζητήσουμε και αργότερα. Είναι επίσης καθήκον μου να ενημερώσω όλους και τους και εισηγητές ότι υπάρχουν τροπολογίες που θα αποσυρθούν και θα ενημερώσω για το ποιες θα είναι αυτές ποια θα είναι η τελική μορφή που θα λάβει το κείμενο και φυσικά τις επόμενες μέρες είμαι στη διάθεσή σας να συναντηθούμε, να το συζητήσουμε, να σας ενημερώσω για οτιδήποτε χρειάζεστε. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπα-Νικολάου. Το επόμενο θέμα τώρα Βλέπετε για τις 9 και 45 και θα πρέπει να περιμένουμε τους συναδέλφους μας και γι' αυτό θα πρέπει να διακόψω τώρα τη συνεδρίαση για λίγα λεπτά. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε ψηφοφορίες αν δεν σεβαστούμε ακριβώς το

So let's continue. Συνεχίζουμε. με την ψηφοφορία για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών με εισηγητή τον κύριο Κορνέλης Ντεγιόγκ. Τροπολογία 1. Υπέρ. Α, συγγνώμη, είναι κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Χες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά θα το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά, γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά. Λοιπόν, τροπολογία 2 ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Είπα τροπολογία 2. Έληξε. Ισοψηφία 12-12. Α, ναι, καλά. Επανάληψη. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 2 ηλεκτρονικά και με τα κουμπιά. Έληξε. 14 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ Κατά. Α, τι δύσκολα που είναι. Πάλι επαλήθευση ηλεκτρονικά. Μα έρχεται. Ψηφίστε ρε παιδιά. Έληξε. 13 υπέρ, 15 κατά. Απορρίπτεται. 4 υπέρ. κατά εποχές επαλήθευση ηλεκτρονικά έληξε 12 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά θα επαληθεύσω 5 έρχεται έληξε 15 υπέρ 14 ε, κατά εγκρίνεται 6 υπέρ θα επιτρέψουμε να ξαναψηφίσουμε την 5 για την κυρία Λάτφορντ. Δέχεστε. Καλά, άρχεται η ψηφοφορία ξανά για την τροπολογία 5 για την κυρία Λάτφορντ. Έληξε. 15-15. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά εποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ κατά ποιες επαλήθευση για την 8 8 14 υπέρ 16 κατά απορρίπτεται συμβιβαστική 1 υπέρ κατά ποιες εγκρίνεται εννέα υπέρ κατά επαλήθευση. Μάχη την ψηφοφορία για την εννέα ηλεκτρονικά. εννέα έλειψη 16 υπέρ 14 ε, κατά εγκρίνεται. 10 υπέρ. Τι θέλετε κύριε Λουά. Δεν συμφωνώ που ξαναψηφίσαμε την 5 και παρακαλώ να δεχτείτε την πρώτη ψηφοφορία μόνο. Γιατί αν είναι έτσι να τις ξαναψηφίσουμε όλες. Δεν γίνεται έτσι, δεν είναι αυτή η συνήθεια. Ζητώ λοιπόν την πρώτη ψηφοφορία να εγκρίνεται. Ευχαριστούμε κύριε Λούαν, αλλά ρώτησα αν συμφωνούν οι συνάδελφοι και συνεφώνησαν. Ναι, ρωτήσατε αλλά όχι όλους, γιατί δεν συμφωνούσαμε όλοι να επαναληφθεί η ψηφοφορία επειδή κάποιος μπήκε στην αίθουσα Μα η κυρία Λάτφορντ ήταν στην αίθουσα, αλλά δεν είχε χρησιμοποιήσει την κάρτα της. Και γι' αυτό, για να είναι σαφή τα πράγματα, θα ζητήσω να ψηφίσουμε αν δέχεστε την επανάληψη που έγινε της ψηφοφορίας για την 5. Ψηφίζουμε λοιπόν συμφωνείτε που επαναλάβαμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 5. Ψηφίζουμε λοιπόν το αν θα λάβουμε υπόψη μας το πρώτο ή το δεύτερο αποτέλεσμα. Όχι. Ψηφίζουμε αν συμφωνούμε να ξανακάνουμε την ψηφοφορία για την πέντε. Καλά. Εάν συμφωνείτε να ξαναψηφίσουμε τώρα Μα εδώ υπάρχει κίνδυνος συγχύσεως. Να ρωτήσετε, δέχεστε το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας όπου είχα ψηφίσει και εγώ. Αυτό να ρωτήσετε. Δεχόμαστε το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας. Αλλιώς θα υπάρξει σύγχυση. Δέχεστε δηλαδή αυτό που αποφασίσατε ότι ξαναψηφίσαμε Ωραία, ερωτώ λοιπόν. Επιβεβαιώνουμε την απόφαση μου που ξανα, κατά την οποία ξαναψηφίσαμε την τροπολογία 5. Όχι, αυτό θα δημιουργήσει σύγχυση. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Λάτφορντ να ρωτήσουμε αν θα λάβουμε υπόψη μας το πρώτο ή το δεύτερο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το αποτέλεσμα της πρώτης ή της δεύτερης ψηφοφορίας. Κύριε Λούαν. Εγώ ρώτησα και οι περισσότεροι δέχτηκαν, δεν ζήτησαν να το ψηφίσουμε ηλεκτρονικά βέβαια, αλλά η πλειοψηφία είχε συμφωνήσει να επαναληφθεί η ψηφοφορία για την 5. Όχι, δεν συνεφώνησαν όλοι. Καλά κύριε Λούαν μου, τότε ερωτώ επιβεβαιώνετε την απόφαση μου σύμφωνα με την οποία ξαναψηφίσαμε όχι με συγχωρείτε η απόφασή σας και το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας γιατί αλλιώς νομίζουν ότι ρωτάτε αν θα ξαναψηφίσουμε τώρα όχι ρωτάτε αν θα δεχτούμε το αποτέλεσμα της δεύτερης ψηφοφορίας ή της πρώτης ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ε, κυρία Πρόεδρε. Ε, είναι, δημιουργήθηκε μία σύγχυση. Υπήρξε η πρώτη ψηφοφορία, μετά ήρθε πράγματι η κυρία Λάτφορντ, ζήτησε να ψηφίσει με την κάρτα της, επαναλάβαμε την ψηφοφορία. Συχνά συμβαίνει αυτό. Απ' την άλλη δεν θέλουμε να έχουμε επαναλήψει συνεχώς γιατί αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Μπορούμε να ψηφίσουμε παρακαλώ επί της τροπολογίας 5 ναι. για να ξεκαθαρίσει το θέμα. Μία τελευταία ψηφοφορία για το άρθρο 5. Θα συμφωνήσετε μαζί μου συνάδελφοι να επαναληφθεί η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 5 αυτό. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι συμφωνείτε. Θα επαναλάβουμε λοιπόν την ψηφοφορία, ηλεκτρονική θα είναι η ψηφοφορία αυτή, για την τροπολογία 5 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας 16 υπέρ 17 κατά <clears throat> απορρίπτεται λοιπόν η πρόταση Επιστρέφουμε λοιπόν στην τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 10. The vote is closed. 17 in favor. 17 υπέρ, 13 κατά, 3 αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε μάλλον ηλεκτρονικά για να είναι ξεκάθαρο το αποτέλεσμα για την 12. Στι της ψηφοφορίας. 17 υπέρ 16 κατά γίνεται δεκτή. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος λοιπόν για την τροπολογία 14. Ψηφίζεται ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, 19 κατά απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά. Αποχές, δεκτό. 16 υπέρ, κατά. Αποχές, γίνεται δεκτή. 17 υπέρ, κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα το τροποποιημένο κείμενο, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα στις ψηφοφορίες, 30 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή, συγχαρητήρια στον εισηγήτη. Πηγαίνουμε στο σημείο 14, τροποποίηση της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για την απλούστευση των θεωρήσεων. Η συγητής είναι ο κύριος Μωράες. Έχει πρώτα το λόγο ο κύριος Μωράες και μετά οι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο. Ευχαριστώ Κίνγκα. Παρά το θόρυβο θα συνεχίσω. Μην ανησυχείς. Θα συνεχίσω. Περιμένετε ένα λεπτό, λέει η πρόεδρος. Μέχρι να φύγουν οι συνάδελφοι που πρέπει να φύγουν. Συνάδελφοι, παρακαλώ, θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Αν θέλετε να φύγετε, φύγετε. Ή μείνετε στην αίθουσα, αλλά αν μείνετε, καθίστε. Okay. Mr. Moraes. Κύριε Μωράης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Κίνγκα. Να κάνω μία σύντομη παρέμβαση για αυτήν εδώ τη συμφωνία και θα εστιάσω στα σημαντικότερα. Η συμφωνία αυτή τροποποιεί την ισχύουσα συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ουκρανία για τη διευκόλυνση χορήγησης θεωρήσεων σε Ουκρανούς πολίτες. Η αρχική συμφωνία είναι σε ισχύ από το 2008 και ο σκοπός της είναι να διευκολύνει τις θεωρήσεις για παραμονή όχι μεγαλύτερη των 9 ημερών μέχρι 180 μέρες για Ουκρανούς πολίτες. Συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαιρούνται από απαιτήσει θεώρησης από το 2005 όταν ταξιδεύουν στην Ουκρανία. Και αυτή η, συμφορία, η συμφωνία συμπεριλαμβάνει συστάσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν ανάμεσα στο Συμβούλιο, των Κομισιόν και την Ουκρανία. Το τελικό κείμενο βασίζεται στην αρχική συμφωνία και τώρα εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το εγκρίνουμε ή όχι. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα μερικών βασικών τροποποιήσεων που έγιναν στην συμφωνία. Το είπα και στις προηγούμενες συζητήσεις μας. ότι οι τροποποιήσεις απλουστεύουν στην ουσία τις απαιτήσει χορήγηση θεώρησης όσον αφορά τον σκοπό του ταξιδιού. Καταργεί το, την εισφορά των 70 ευρώ για την χορήγηση. Απλοποιεί τη διαδικασία θεώρησης για πολλαπλές εισόδους στη χώρα, διαδοχικές εισόδους. Επίσης αναφέρεται στην διαδικασία εισόδου με τα βιομετρικά διαβατήρια. Το συζητήσαμε και σε προηγούμενη ολομέλεια και λόγω της πολιτικής κατάστασης στην Ουκρανία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκφράσει τις ανησυχίες της ιδιαίτερα όσον αφορά την αποτυχία της Ουκρανίας να εφαρμόσει πλήρως όλα όσα είχαν συμφωνηθεί στο Σύμφωνο Οικονομικής Συνεργασίας Γι' αυτό θεωρώ πως η τροποποιημένη συμφωνία είναι σημαντικό βήμα προ τα εμπρός. Και κυρία Πρόεδρε, μπορούμε να συζητήσουμε την ε, πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία και αν έχει ε, υπάρξει πρόοδος και το θεωρώ ε, σημαντικό. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψη των συναδέλφων σήμερα για την κατάσταση στην Ουκρανία. Θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να πω ότι προθεσμία για τροπολογίες είναι 5 Φεβρουαρίου Η γνωμοδότηση υιοθετήθηκε στις 22 Ιανουαρίου και αναμένω τα σχόλιά σας. Κύριε Μωρές, ευχαριστούμε. Η κυρία Μπένοκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Η δική μας ομάδα συμφωνεί με τα συμπεράσματα της έκθεσης και συμφωνούμε με την τροποποιημένη αυτή συμφωνία. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ε, τροποποιήσεις για τη διευκόλυνση έκδοσης θεώρησης, για τις χώρες αυτές της ε, Ανατολικής Ευρώπης, θεωρώ πως είναι καλό να εναρμονίσουμε γενικότερα τις διατάξεις για όλες αυτές τις χώρες. Αυτά από εμάς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ποτάσοβιτς, εκ μέρους του ΕΛΚ, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είμαστε υπέρ της συμφωνίας αυτής, όπως ανέφερε και ο κύριος Μωράες, Ακόμα και αν η πολιτική κατάσταση στην Ουκρανία έχει υπάρξει αντικείμενο επικρίσεων, αυτό δεν είναι κάτι που θα πρέπει να επηρεάσει τη διευκόλυνση των Ουκρανών πολιτών να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες όπως ε, θρησκευτικές ομάδες, δημοσιογράφοι, νέοι, μέλη της, ε, των χωρών Ανατολικής Συνεργασίας και στην Επιτροπή αυτή εδώ και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων υπάρχει η τάση να συνενέσουμε στην τροποποίηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ποτασιεβίτς. Το λόγο έχει η Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Είμαι Αντιπρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Χορήγησης Θεωρήσεων. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την θετική του έκθεση. Να ευχαριστήσω και τους ευρωβουλευτές που μόλις τώρα εξέφρασαν την στήριξή τους στη συμφωνία αυτή. Ο κύριος Μωράς, πιστεύω, συνοψίζοντας μας έδωσε μία εικόνα του πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία. Επιτρέψτε μου να κάνω ορισμένες πρόσθετε παρατηρήσει όμως. Πράγματι υπάρχει ήδη μία συμφωνία με την Ουκρανία για θεωρήσει από την 1η Ιανουαρίου 2008. Και σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε ότι η αρχική συμφωνία ήδη έχει προσκομίσει πολλά ωφέλη στην Ουκρανία και θα σας δώσω και μερικά παραδείγματα από το 2009 και το 2011 ο αριθμός των θεωρήσεων που χορηγήθηκαν στην Ουκρανία αυξήθηκε κατά 33,8%. Και ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των θεωρήσεων που χορηγήθηκαν πάνω από το 1 τρίτο χορηγήθηκαν με συνοπτικέ διαδικασίε και υπήρχε με, ε, πολύ μικρό ποσοστό άρνηση έκδοσης θεωρηση. Πιστεύω ότι γενικότερα ο πληθυσμό της Ουκρανίας θα ωφεληθεί και πιστεύουμε ότι η τροποποίηση του κανονισμού θα ωφελήσει εν γέννη τους Ουκρανούς. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε πολύ υπέρ της γρήγορη. κύρωση της συμφωνίας και να σας πω επίσης ότι η τροποποίηση της συμφωνίας που έχουμε της αντίστοιχη με τη Μολδαβία θα πρέπει και εκείνη να ολοκληρωθεί σύντομα. Δεν θα θέλαμε να δούμε καθυστερήσεις στη συμφωνία με τη Μολδαβία, διότι υπάρχει το ενδεχόμενο η πλευρά της Μολδαβίας να ερμηνεύσει αυτή την καθυστέρηση πολιτικά. Ξέρω ότι είναι στην ημερήσια διαταξή σας, στα προσεχώς, η συζήτηση για τη συμφωνία με τη Μολδαβία, όμως θα ήθελα να σας παρακαλέσω να γίνει αυτό σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Επιστρέφω τώρα στον εισηγητή. Έχει το λόγο ο κ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που συμφωνούν ότι και στην αιτιολογική έκθεση ότι η περίπτωση αυτή συνιστά μια πολιτική ενθάρρυνση προς την Ουκρανία και στους κατοίκους της, στους πολίτες της Ουκρανίας για να υπάρξει πολιτική πρόοδος. Οι διευκολύνσεις για τις θεωρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν και γι' αυτό το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμφωνήσει με την πρόταση αυτή. Και ευχαριστώ τους Σκιώδης για τη συμφωνία τους. Ευχαριστώ κύριε Μωράης. Τώρα συνεχίζουμε. Περνάμε τώρα στο δεύτερο θέμα σχετικά με τις θεωρήσεις πρόκειται για την έκθεση που αφορά ε, την τροποποίηση των καταλόγων ε, που, των χωρών που υπόκεινται σε ε, θεωρήσεις για την περιοχή Σέγγεν. Υπάρχει και η έκθεση μέρα για το ίδιο θέμα. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον εκπρόσωπο ε, της Επιτροπής και μετά στην κυρία Γκαμπριέλ. Και θα δώσω και το λόγο στην Ιρλανδική Προεδρία εφόσον επιθυμούν να παρέμβουν. Το λόγο έχει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Και εγώ θα, και το θέμα αυτό θα το παρουσιάσω εγώ και ο κύριος Ντεκόστερ θα παρουσιάσει τα δύο επόμενα θέματα για τις θεωρήσεις. Υπάρχει μια πρόταση λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροποποίηση του κανονισμού 539. Έχετε απολύτως δίκιο που μας υπενθυμίζετε και υπενθυμίσατε στα μέλη ότι υπάρχει και μια άλλη τροπολόγηση της 539 υποσυζήτηση στα πλαίσια της μορφής συνεργασίας ανάμεσα στους συνομοθέτες. Δεν πρέπει να αναμειγνύουμε τα δύο. Αυτή την οποία εξετάζουμε σήμερα είναι η τακτική αναθεώρηση από πλευράς Επιτροπής ε, των παραρτημάτων και των καταλόγων του 539 σχετικά με τον κατάλογο των χωρών οι οποίες υπόκεινται σε θεωρήσεις και αυτών οι οποίες είναι ελεύθερες θεωρήσεων για να έρχονται οι πολίτες τους στην περιοχή Σέγγεν, στη ζώνη Σέγγεν. Έχει ήδη αναθεωρηθεί ο 539 από το 2001 8 ή 9 φορές. Η τελευταία αναθεώρηση έγινε το 2010 όταν ε, μετακινήθηκαν στις θετικούς λεγόμενους καταλόγους κάποιες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και επίσης ε, η Ταϊβάν. Η αναθεώρηση αυτή όπως είπα γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά περίπτωση εξετάζουμε τις προτάσεις ε, και τις συστάσεις ε, των χωρών μελών για τις ε, μεταφορές χωρών από την ένα κατάλογο στον άλλο. Ελέγχονται επίσης και τα κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός 539. Ίσως και να είναι η τελευταία αναθεώρηση γιατί στο μέλλον θα λαμβάνουμε υπόψη μας και διαφορετικά κριτήρια αλλά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα συζητήσετε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Προς στιγμή εμείς εργαζόμεθα επί τη βάση των, των κριτηρίων που υπάρχουν τώρα εξετάζουμε τους κινδύνους ε, άτακτων μορφών ε, μετανάστευσης, απειλών στην εθνική ασφάλεια και στη δημόσια ασφάλεια και το θέμα των εξωτερικών σχέσεων γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, κάτι το οποίο έχει σχέση με την συνοχή στην αντιμετώπιση της περιφέρειας από την οποία προέρχεται η χώρα. Είδαμε ποιες ήταν οι δυνατότητες λοιπόν μετακίνησης από τον ένα κατάλογο στον άλλο και μετά από προσεκτική εξέταση των προτάσεων των κρατών μελών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι χώρες οι οποίες αναφέρονται στην πρόταση θα πρέπει να μεταφερθούν στη θετική λίστα Κανένα κράτος μέλος δεν πρότεινε τη μετακίνηση χώρας στην αρνητική λίστα, στον αρνητικό κατάλογο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, γιατί παρόλα αυτά ε, σε σχέση με ορισμένες χώρες ε, που είναι ελεύθερες θεωρήσεων κάποια προβλήματα ναι. υπάρχουν. Αλλά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία θα προτείνουν τις πιθανές μεταφορές. Οι χώρες λοιπόν τις οποίες προτείνουμε τώρα αναφέρονται είναι μικρές βασικά χώρες της Καραϊβικής και χώρες νήσι του Ειρηνικού, δεν θα αναφερθώ σε όλες τις χώρες. 16 μικρές χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο και μια τρίτη κατηγορία είναι μια ειδική κατηγορία Βρετανών πολιτών οι οποίοι υπόκεινται σε διαφορετικές νομικές υποχρεώσεις και δικαιοδοσίες και θα πρέπει να μετακινηθούν και αυτοί στον θετικό κατάλογο. Τέλος, και για να μπει στα πρακτικά να πω ότι σύμφωνα με την πρόταση αυτή θα συμπεριλάβουμε στην αρνητικό κατάλογο και το, το Νότιο Σουδάν. Επειδή το Σουδάν είναι έτσι και αλλιώ στον αρνητικό κατάλογο, το Νότιο Σουδάν σαν τμήμα του πρέπει να παραμείνει και αυτό εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η πρόταση της Επιτροπής. Να πω επίσης ότι ορισμένες άλλες χώρες έγιναν αντικείμενο αναφοράς από τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν και πιέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρόλα αυτά θεωρεί ότι σε αυτή τη φάση δεν θα πρέπει να μεταφερθούν οι χώρες αυτές στον θετικό κατάλογο αλλά σε μελλοντικές μεταρρυθμίσεις ε, το θέμα τους θα εξεταστεί. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δώσατε να παρουσιάσω αυτή την σοβαρή πρόταση της Επιτροπής. Ευχαριστώ η συγγήτρια κυρία Γκαμπριέλ. Ευχαριστώ πρόεδρε να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας παρουσίασε το πλαίσιο και το περιεχόμενο του κανονισμού σε μια πρώτη φάση να επανέλθω σε κάποια από τα κομβικά στοιχεία του περιεχομένου και να προσπαθήσουμε να έχουμε και κάποιες συμπληρωματικές διευκρινήσεις από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με αυτό που είπε η Επιτροπή, ότι πρόκειται για μια έκθεση η οποία ίσως να είναι η τελευταία της σειράς. Ε, πρόκειται δηλαδή για μια έκθεση ελέγχου συνέχειας αν θέλετε. Υπάρχουν κάποιοι κατάλογοι οι οποίοι ισχύουν και υπάρχει δυνατότητα για πολίτες ορισμένων χωρών να περάσουν στους θετικούς καταλόγους. Είναι σαφές ότι τα κριτήρια όπως η παράνομη μετανάστευση, η ασφάλεια ε, και οι εξωτερικές ε, σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και μπορούν τα κριτήρια αυτά να μας επιτρέψουν να μιλήσουμε ανοιχτά για τρεις κατηγορίες χωρών. Πρώτη κατηγορία είναι οι 16 χώρες του Ειρηνικού και η δεύτερη κατηγορία οι λεγόμενοι Βρετανοί πολίτες και τέλος το Νότιο Σουδάν. Εδώ θα ήθελα να θέσω ορισμένες ερωτήσεις. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να μας δώσει αριθμούς. Ε, τι πληθυσμός είναι αυτός ο οποίος καλύπτεται από τον κανονισμό αυτό και για τους Βρετανούς πολίτες ε, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Δεύτερον, θα έχουμε και πληροφορίες σχετικά με το πόσες χώρες έχουν ε, ε, προξενικές αντιπροσωπείες στις χώρες αυτές και κατά πόσον η αλλαγή αυτή θα διευκολύνει την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και να επιμείνω και στην αρχή της αναλογικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν κατάλαβα καλά στην έκθεση αυτή, η εξαίρεση της υποχρέωσης έκδοσης θεωρήσεων για τους πολίτες των χωρών αυτών θα τεθεί σε λειτουργία τη στιγμή που θα υπογραφεί μια διμερή συμφωνία ανάμεσα στις χώρες αυτές και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν υπάρχει δηλαδή ομαδική διαπραγμάτευση αλλά κατά περίπτωση, κατά χώρα. Αυτά. Τελειώνοντας θα ήθελα για μια ακόμη φορά να εκφράσω την ικανοποίησή μου γιατί ο διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ιδιαίτερος παραγωγικός και ελπίζω με το, το ταχύτερο δυνατόν με το Συμβούλιο να κάνουμε τα απαιτούμενα βήματα. Ευχαριστώ κυρία Γκαμπριέλ. Δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Α, υπάρχει η κυρία Σντάνοκα που έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνο και εγώ, συμφωνεί και η ομάδα μας. Είναι θετικό να μεταφέρεται ένα κράτος από την αρνητική λίστα στη θετική. και 16 ήταν αυτά τα κράτη που μετακινήθηκαν. Αυτό που με απασχολεί είναι οι Βρετανοί πολίτες. Είχαμε ήδη τροποποιήσει τον κανονισμό. Και μπορείτε να μας εξηγήσετε περισσότερο τι γίνεται με τις κατηγορίες αυτές, Ποιου αφορούσε η προηγούμενη τροποποίηση, ποιου τώρα, αν υπάρχει κάποια κατηγορία που δεν καλύπτεται από τη δική σας πρόταση ή αν τα έχετε καλύψει όλα. Και συμπεριλαμβάνονται όλοι οι Βρετανοί πολίτες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντανόκα, κύριος Μίσα. Μάλιστα κυρία μου, και εγώ τα ίδια ερωτήματα έχω με την κυρία Γκαμπριέλ. Μια αποσαφήνιση θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια. Στο επίπεδο των αρχών συμφωνούμε, η κατάργηση των θεωρήσεων θα διευκόλυνε πολλούς φοιτητά, φοιτητρια και άλλους. Αλλά και η πρόταση κανονισμού λέει ότι οι ενδιαφερόμενες χώρες δεν αποτελούν κανέναν κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης ή διατάραξης της τάξεως. Οι δε ενωσιακοί πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν τις χώρες αυτές επίσης δεν θέτουν πρόβλημα. Υπάρχει βέβαια μια ειδική κατηγορία των υπερποντίων Βρετανών πολιτών που απολαμβάνουν και αυτή την ελεύθερη διακίνηση στο χώρο Σέγγεν. Συνδεχόμαστε και αυτή την πρόταση της κυρίας Γκαμπριέλ και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να εγκρίνει σύντομα. Βατκόσκι. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ολοκληρώσαμε τις συζητήσεις για αυτό το σημείο. Ωστόσο υπάρχει πρόταση να καταργηθούν οι θεωρήσεις για ορισμένους Βρετανούς πολίτες. Μία ερώτηση έχω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γίνεται να εξαιρεθούν ορισμένοι Ουκρανοί πολίτε από τι απαιτήσει ε, θεώρηση. Έχουμε καταργήσει κάποιε ε, κάποιες εισφορές, όμως πιστεύω πως οι Ουκρανοί πολίτες έχουν το δικαίωμα να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεώρηση. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Ας αρχίσω από την τελευταία. Εάν μπορούμε να εξαιρέσουμε και τους Ουκρανούς πολίτες. Φοβάμαι ότι δεν είναι αυτός ο σκοπός της παρούσης πρότασης. Όπως ίσως γνωρίζετε, υπάρχει ένας διάλογος με την Ουκρανία για τις θεωρήσεις, ο οποίος κάποια στιγμή θα οδηγήσει στην κατάργηση της ε, απέτηση σε θεώρησης για την Ουκρανία. Αυτή τη στιγμή συζητούμε με την Ουκρανική πλευρά για αυτό το ζήτημα. Δεν μπορώ όμως να σας πω ακριβώς πότε αυτό θα υλοποιηθεί, αλλά να σας πω ότι ο διάλογος συνεχίζεται και θα καρποφορήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τώρα, Μία από τις ερωτήσεις που μου κάνατε ήταν βασισμένη στην πρόταση της Επιτροπής για πόσους ακριβώς ανθρώπους μιλάμε. Λοιπόν, τα νούμερα τα έχω μπροστά μου. Συνολικά αναφερόμαστε σε νησιά κράτη στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό έχουμε να κάνουμε με περίπου λίγο πάνω από 4 εκατομμύρια ανθρώπους και όσον αφορά τους υπερπόντους Βρετανούς είναι ακόμα 300.000. Στο σύνολό της η πρόταση αυτή αφορά 4,5 εκατομμύρια λοιπόν ανθρώπους. Τώρα για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Όπως ξέρετε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει ένα αρκετά περίπλοκο σύστημα πολιτών με διαφορετικά δικαιώματα. Είναι περίπλοκο το ποιος είναι Βρετανός πολίτης και πόσο. Στο παρελθόν μεταφέραμε αρκετές κατηγορίες ε, υπερπόντιων Βρετανών από τον αρνητικό στον θετικό κατάλογο. Και τώρα προτείναμε να μεταφερθούν και οι υπόλοιποι. Το βρετανικό λοιπόν σύστημα τους ονομάζει Βρετανούς πολίτες από τις υπερπόντιες περιοχές. Είναι υπήκοοι του στέματος. Έχ, ορισμένοι έχουν το δικαίωμα ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορισμένοι όχι, όμως σε γενικές γραμμές βασισμένοι στις αξιολογήσεις μας, αυτοί οι πολίτες δεν αποτελούν κίνδυνο για παράνομη μετανάστευση. έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα που ανταποκρίνονται στα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου. Για τους λόγους αυτούς λοιπόν δεν θεωρούμε ότι θα προκαλέσουν κάποια προβλήματα όσον αφορά τα κριτήρια που ανέφερα. Επίσης, άλλη μία ερώτηση, αν δεν κάνω λάθος, είναι για την προξενική κάλυψη στα νησιά αυτά. Και αυτός ίσως είναι και ένας άλλος λόγος να τους μεταφέρουμε στον θετικό κατάλογο, διότι σε γενικές γραμμές η προξενική κάλυψη σε αυτά τα νησιά τόσο στην Καραϊβική όσο στον και στον Ειρηνικό είναι ατελής, δεν είναι παρκής. Πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να ταξιδέψουν πολύ μακριά για να πάρουν βίζα. Να σας δώσω παραδείγματα. Στα νησιά του Ειρηνικού, για παράδειγμα, Υπάρχουν μόνο δύο κράτη-μέλη που έχουν προξενικές αρχές. Η Πορτογαλία στο Ανατολικό Τιμόρ και η Γαλλία στο Βανουάτου. Τι σημαίνει αυτό, ότι όλα τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν καμία προξενική αντιπροσωπεία κράτους μέλους της, Ευρωπαϊκού, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό κάποιος που, που μένει στα νησιά Μάρσαλ πρέπει να ταξιδέψει πολλά χιλιόμετρα στα νησιά Βανουάτου για να πάρει μια βίζα. Στην Καρεβική η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη, όμως και εκεί δεν υπάρχει επαρκής προξενική κάλυψη. Και η προξενική κάλυψη που υπάρχει είναι βασισμένη στους ιστορικούς δεσμούς των χωρών αυτών με τα κράτη-μέλη. Ο τώρα, αμοιβαιότητα. Έχετε δίκιο. Πρέπει να διασφαλίσουμε την αμοιβαιότητα. Γι' αυτό λοιπόν η άρση σε υποχρεώσεις θεώρησης βρίσκονται σε στάδιο διαπραγματεύσεων και επιθυμούμε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών. Και φυσικά κατά τη διάρκεια των συζητήσεων θα προσπαθήσουμε να διασφαλιστεί η αρχή της αμοιβαιότητας. Νομίζω πως απάντησα στις ερωτήσεις σας και αν έχω παραλείψει κάτι, παρακαλώ πείτε μου. Νομίζω όμως πως σας κάλυψα. Η ε, κυρία Ντανόκα βλέπω θέλει κάτι να ρωτήσει, λέει η πρόεδρος. Ναι, με συγχωρείτε, δεν απαντήσατε στην δική μου ερώτηση. Για τις κατηγορίες των Βρετανών, υπερπόντι, Βρετανοί, Βρετανοί, θα μας καλύψει ο κανονισμός αυτός. Ναι, με συγχωρείτε. Ναι. Εάν μετακινήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, όπως προτείνουμε, στον θετικό κατάλογο, τότε δεν υπάρχει κανένας άλλος Βρετανός πολίτης ή κατηγορία Βρετανού πολίτη που θα βρίσκεται εκτός πεδίου του κανονισμού. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό βήμα όσον αφορά τους Βρετανούς πολίτες. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Γκάμπριελ, θα ζητήσω από την Ιρλανδική Προεδρία να παρέμβουν και να μας πούν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο Συμβούλιο. Κύριε Ράιαν, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που είχα την ευκαιρία να έρθω εδώ και να σας μιλήσω γι' αυτό. Άκουσα την εισηγήτρια και τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Έλαβα υπόψη τις ερωτήσεις τους και τις απαντήσεις της Επιτροπής. Να σας δώσω τώρα πληροφορίες για τις νεότερες εξελίξεις στο Συμβούλιο και να σας πω τι σκοπεύουμε εμείς να κάνουμε. Αυτός ο κανονισμός για τις θεωρήσεις παρουσιάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις 27 Νοεμβρίου του περασμένου έτους. Διεξήχθησαν συζητήσεις σε υπουργικό επίπεδο τον Δεκέμβριο του 2012. Η πρώτη πρόταση υποβλήθηκε τέλη Ιανουαρίου στην ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις. Γενικά έγινε αποδεκτή από τα κράτη-μέλη θετικά, δεν υπήρξε κανένα κράτος μέλος που επιθύμησε να μεταφέρει από τον θετικό στον αρνητικό κατάλογο κάποια χώρα. Αναφέρθηκαν όμως κάποιες ε, αμφιβολίες σχετικά με τρία κράτη-μέλη, αλλά ελπίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι μεγάλο πρόβλημα για τις εξελίξεις. Τώρα, όπως ανέφερε και η Κομισιόν, πολλά κράτη-μέλη πρότειναν την εισαγωγή των 16 αυτών κρατών στον θετικό κατάλογο. Κάποια κράτη-μέλη όμως εξέφρασαν τις ανησυχίες τους και τις ανησυχίες τους επίσης και για το ζήτημα της συνοχής. Στις 22 Φεβρουαρίου θα συνεδριάσει η ομάδα εργασίας για τις θεωρήσεις και εμείς ως Ιρλανδική Προεδρία έχουμε στόχο να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για αυτό το συντομότερο δυνατόν. Γι' αυτό ελπίζουμε σε καλή συνεργασία και στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ράιεν. Το λόγο έχει η συγχύτρια. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το σχόλιο μου θα είναι πάρα πολύ σύντομο. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν μέρος στη συζήτηση. Ευχαριστώ την Επιτροπή και την Ιρλανδική Προεδρία που μας έδωσε κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες έτσι ώστε να κατανοήσουμε σε βάθος το θέμα. Να τους ευχαριστήσω επίσης και για τον διάλογο ο οποίος έχει ήδη αρχίσει να λειτουργεί. Όπως το είπε και η Ιρλανδική Προεδρία, ελπίζω το ταχύτερο δυνατόν να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα περνάμε στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης από κοινού συζήτηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής ε, για την ε, ανάπτυξη της πολιτικής χορήγησης θεωρήσεων και για την λειτουργία της επιτόπιας συνεργασίας Σέγγεν κατά τα πρώτα δύο χρόνια ε, της εφαρμογής του κώδικα θεωρήσεων. Ο κ. Ντεκόστερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Βάζοντας τα δύο αυτά θέματα στην ημερήσια διάταξη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ακολούθησε τη λογική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν στις 7 Δεκεμβρίου υιοθέτησε το λεγόμενο πακέτο για τις θεωρήσεις με τρία βασικά χαρακτηριστικά, την τροπολόγηση των θεμάτων που ήδη συζητήσατε, αλλά και την ανακοίνωση προς το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη της πολιτικής των θεωρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ανάπτυξη των επιτόπιων συνεργασιών στα πλαίσια του Σέγγεν. Ανάμεσα σε αυτά τα τρία στοιχεία υπάρχει μια κάποια λογική. Εγώ παρουσιάζω τα δύο πρώτα από κοινού, αν και η φύση των δύο στοιχείων μπορεί να είναι λίγο διαφορετική. Η ανακοίνωση στην ουσία είναι μια ανακοίνωση πολιτικών θέσεων. Εκφράζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περαιτέρω ε, προσπάθειες ανάπτυξης της κοινή πολιτικής των θεωρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι σε εύθετο χρόνο θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή στο σύστημα αυτό. Η έκθεση είναι μια προσπάθεια αξιολόγησης, αν θέλετε, της προσπάθειας που έχει γίνει ε, στο πλαίσιο της επιτόπιας συνεργασίας Σέγγεν κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του κώδικα θεωρήσεων. Να ξεκινήσω με την ανακοίνωση λοιπόν ε, την πολιτική αν θέλετε. Δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε από το πουθενά. Υπάρχει ένα σαφέστατο θέμα στον τομέα της πολιτικής των θεωρήσεων με τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με τον οικονομικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά από ευρήματα στα πλαίσια και των εργασιών του ομάδα των 20 και στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας. Έχει εξετάσει γενικά τις πιθανές εξελίξεις στον τομέα αυτό στον τομέα επίσης της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει ένας τομέας στον οποίο υπάρχουν δυνατότητες για περαιτέρω εξελίξεις που μπορεί να οδηγήσουν σε οικονομική ανάπτυξη και σε δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Στο παρελθόν, αναπτύσσοντας την πολιτική των θεωρήσεων, θεωρούσαμε εμείς ότι είναι ένα απλό συνοδευτικό μέτρο αν θέλετε του τομέα Σέγγεν εμένοντας κυρίως τα θέματα ασφάλειας. Αλλά υπάρχει και μια διάσταση ελευθερίας αν θέλετε. Με ποια έννοια. Να υπενθυμίσω εδώ κάποια από τα στοιχεία τα οποία έχουν σημασία. Ένα από τα βασικά κεκτημένα του Σέγγεν είναι ότι με μία θεώρηση μπορεί να επισκεφθεί κανείς και τις 26 χώρες της Ένωσης που συνιστούν το Σέγγεν. Ενώ παλαιά χρειαζόταν κανείς μία διαφορετική θεώρηση για κάθε μία από τις χώρες που ήθελε να επισκεφθεί. Η ομάδα των 20 πρότεινε, το G20 πρότεινε λοιπόν αυτού του είδους την περιφερειακή αντίληψη για τη χορήγηση των θεωρήσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει ήδη προσφέρει πολλά. Η πολιτική των θεωρήσεων λοιπόν πράγματι προωθεί την κινητικότητα, αν και πάντα υπάρχουν ορισμένα εμπόδια και θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάποιους αριθμούς Ήδη αναφέρθηκα στην αύξηση του αριθμού των θεωρήσεων, των αιτήσεων συγγνώμη, για θεωρήσεις. Ανάμεσα στο 2009 και στο 2011 υπήρξε μια αύξηση αιτήσεων κατά 32%. Ένα τρίτο επιπλέον δηλαδή αιτήσεων και με ένα ποσοστό άρνησης χορήγησης που δεν ξεπερνά κατά μέσο όρο το 5,5%. Η συμφωνία λοιπόν του 2010 σαφώς και έχει ε, διευκολύνει την χορήγηση των θεωρήσεων. Θα πρέπει όμως να σταθούμε πιο προσεκτικά στο τι ε, στο μέλλον, στο ποιες θα είναι οι οικονομικές επιπτώσεις. Πώς μπορούμε σαν παράδειγμα να διευκολύνουμε τις διαδικασίες ε, πολιτών που να ταξιδεύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέματα ασφάλειας είναι επίσης θέματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν με την εφαρμογή της κοινή πολιτικής. Όπως είπα, ο, ο ε, κώδικας αυτός θεωρήσεων ήταν ένα είδος επαναστατικών θα έλεγα μέτρων, σειράς μέτρων. Θα δείτε όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέγει ότι υπάρχει ακόμα μεγάλο περιθώριο ε, βελτιώσεων στα πλαίσια της εφαρμογής των συμφωνιών αυτών. Πρώτον λοιπόν σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο θα πρέπει εμείς να έχουμε πάντα υπόψη τις οικονομικές επιπτώσεις και να διευκολύνουμε τις υπάρχουσες, να ε, μάλλον βελτιώσουμε τις υπάρχουσες διευκολύνσεις. Μέσω μακροπρόθεσμα Εξετάζοντας τις συνέπειες των συμφωνιών αυτών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ε, σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις. Και προς την κατεύθυνση αυτή να αναφέρω ότι πριν από το τέλος του ενεστώτος έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανέλθει με μια πλήρη αξιολόγηση της εφαρμογής της συμφωνίας και η αξιολόγηση αυτή θα συνοδευτεί από μία πρόταση η οποία να τροπολογεί το σύνολο των συμφωνιών των επιμέρους. Όπως έχω ήδη πει, η αναθεώρηση αυτή δεν θα έχει μόνο την αντίληψη την οποία πρεσβεύει το Σέγγεν, αλλά θα λαμβάνει υπόψη σαφώς και τις οικονομικές επιπτώσεις αυτών των διαδικασιών που προέρχονται από τις συμφωνίες των θεωρήσεων. Η καλύτερη διευκόλυνση βέβαια είναι η απαλλαγή στη συγκεκριμένη περίπτωση. Η υπάρχουσα πρόταση, η οποία είναι υποσυζήτηση, εμπνέεται πάντα από την παλαιότερη θα έλεγα παραδοσιακή αντίληψη για το Σέγγεν. Στο μέλλον, όταν αποφασίσουμε να κάνουμε προτάσεις τροπολόγησης στον κατάλογο, θα λάβουμε υπόψη περισσότερο από ό,τι σήμερα τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις. Η ανακοίνωση αυτή είναι πως πρόεδρε δίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδέες για μελλοντικές προτάσεις έτσι ώστε να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της πολιτικής χορήγησης θεωρήσεων. Είναι ε. μια καλή λοιπόν ευκαιρία για τις συζητήσεις που τις οποίες κάνουμε. Δεν συζητάμε ακόμα κάποια πιο συγκεκριμένα μέτρα, αλλά πρόκειται για μια πολιτική συζήτηση. Η πολιτική συζήτηση αυτή θα πρέπει να ολοκληρωθεί και θα επιτρέψει άμα τη ολοκληρώσει τη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη όλες τις ε, ε, επιπτώσεις στην οικονομία. Δεύτερον, υπάρχει και η έκθεση ε, της Επιτροπής για την Επιτόπια Συνεργασία Σέγγεν. Η επιτόπια συνεργασία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της χορήγησης θεωρήσεων της πολιτικής χορήγησης θεωρήσεων. Έχουμε τους κανόνες που αποφασίζονται από τις Βρυξέλλες, αλλά υπάρχουν τοπικές συνθήκες στις διάφορες περιοχές του κόσμου εντελώς διαφορετικές. Καταρχάς κίνδυνοι στις οποίες εκτίθενται ορισμένες κατηγορίες. Παιδιά από μια χώρα που θέλουν να έρθουν για καλοκαιρινά μαθήματα δεν δημιουργούν προβλήματα δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το χρόνο παραμονής τους. Ενώ σε άλλες χώρες μπορεί να υπάρχει μια τάση κατάχρησης κάποιων διευκολύνσεων έτσι ώστε φοιτητέ ας πούμε να παραμείνουν επιπλέον. Αυτό είναι ένα από τα θέματα το οποίο θα πρέπει να συζητιέται στα πλαίσια των επιτόπιων συνεργασιών. Ποιες επιμέρους κατηγορίες δημιουργούν πρόβλημα. Καταρχάς, ε, τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται. Υπάρχει η Γενική Συμφωνία που προβλέπει ένα κατάλογο εγγράφων, αλλά αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να ορίζονται καλύτερα σε επιτόπιο επίπεδο. Σαν παράδειγμα, πιστοποιητικό απασχόληση σε μία χώρα μπορεί να έχει κανείς ένα κατάλογο όπου, με όπου αριθμούνται αν θέλετε ε, οι προηγούμενοι εργοδότες του υποψηφίου. Ε, σε μια άλλη χώρα έχει κανείς ένα πιστοποιητικό το οποίο δεν προέρχεται από έναν εργοδότη αλλά προέρχεται από μια κρατική υπηρεσία. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ε, μια εναρμονισμένη αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες. Υπάρχουν λοιπόν πολλά να γίνουν στα πλαίσια όλων αυτών των δικαιοδοσιών. Η Συμφωνία για τις Θεωρήσεις λέγει ότι για κάθε δικαιοδοσία θα πρέπει να υπάρχει και ένας κάποιος αριθμός εκθέσεων. Το 2011 όταν ήρθαν οι πρώτες εκθέσεις δεν είχαν ε, τεθεί σε λειτουργία όλες οι επιμέρους επιτόπιες συνεργασίες έγκαινοι. Κάποιες από αυτές είχαν τεθεί σε λειτουργία πάρα πολύ πρόσφατα. Και αυτό μας έκανε να σκεφτούμε για το αν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ε, ε, τις τοπικές αυτές συνεργασίες. Και όταν πήραμε τις επόμενες εκθέσεις για την πρόοδο το 2012, Είδαμε ότι υπήρξε περαιτέρω ενεργοποίηση των επιτόπιων μορφών συνεργασίας και οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να σας πω στην ουσία είναι παράρτημα στην έκθεση που σας υποβάλλουμε τώρα. Έχουν αποσταλεί στον πρόεδρο της Επιτροπής Λίμπε και νομίζω ότι εν τότο για τα δύο χρόνια είχαμε 140 επιμέρους εκθέσεις για επιμέρους επιτόπιες συνεργασίες. Αν θέλετε λοιπόν να γνωρίζετε περισσότερα για το πώς λειτουργεί η πολιτική της χορήγησης θεωρήσεων στις διάφορες χώρες και για το πώς εφαρμόζεται στις διάφορες χώρες, ίσως θα πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά τις εκθέσεις αυτές. Όταν είδαμε τις εκθέσεις αυτές, εμείς προχωρήσαμε με την σύνταξη της παρούσης εκθέσεως, που δεν απαιτείται επίσημα από τη Συμφωνία Σέγγεν, είναι ένα επιμέρο στοιχείο που συνεισφέρει στην πλήρη εφαρμογή. Δεύτερον υπάρχει ανάγκη βελτίωσης και αυτό θα πρέπει να γίνει και μέσω μεμονωμένων συστάσεων προς ε, τα, ε, τα προξενία στις διάφορες χώρες ε, κάποιων επιμέρους μέτρων. Επί τη βάση λοιπόν όλων αυτών των εκθέσεων Έχουμε αναπτύξει κάποιες συστάσεις για όλους τους εμπλεκομένους σε τοπικές μορφές συνεργασίας Schengen. Θα ήθελα εδώ, Πρόεδρε, να σας δώσω κάποιες επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία και τη λειτουργία των επιτοπίων συνεργασιών πριν από τη συμφωνία για τις θεωρήσεις ε, υπεύθυνη ήταν η περιστρεφόμενη προεδρία του Συμβουλίου αλλά με τη νέα συμφωνία για τις θεωρήσεις οι ευθύνε για τον συντονισμό των επιτοπίων συνεργασιών δόθη πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διασφαλιστεί με καλύτερο τρόπο η συνέχεια της λειτουργίας τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εκείνη τη φάση ήταν υπεύθυνη επίσης και για τις ευρωπαϊκές αντιπροσωπίες. Με τη δημιουργία του ΕΑΣ άλλαξαν τα πράγματα αυτά. Δεν είναι τμήματα πλέον των υπηρεσιών της Επιτροπής. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το ΕΑΣ κανένας δεν σκέφτηκε τι σημαίνει αυτό για την ευθύνη της λειτουργίας του συστήματος Schengen και αρχηγοί ε, πολλών γενικά ε, αρχηγών αντιπροσωπιών είπαν ότι δεν αναγνωρίζουν συγκεκριμένη αρμοδιότητα εκεί και ότι αυτά είναι θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δείτε λοιπόν ότι στα πλαίσια των συμπερασμάτων και των ε, συστάσεων οι πρώτες αφορούν ακριβώς τον ρόλο των, των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατευθυντήρια βασική αρχή είναι η κατανομή του βάρους, όχι μόνο ανάμεσα στον ΕΑΣ και της Επιτροπής, αλλά και ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπάρχει η δυνατότητα εκχώρησης ορισμένων αρμοδιοτήτων προς τα κράτη-μέλη. Να προσθέσω εδώ ότι η χρήση ε, των ανθρωπίνων πόρων από το ΕΑΣ και από την Επιτροπή είναι θέματα τα οποία ε, πρέπει να ρυθμιστούν. Δεν είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα βέβαια. Οι αρχηγοί των αντιπροσωπιών κατανοούν στις περισσότερες περιπτώσεις ότι η κινητικότητα είναι ένα όλο και περισσότερο ε, χαρακτηριστικό αν θέλετε των διεθνών μορφών συνεργασίας και οι τοπικές αρχές που ασχολούνται με τα θέματα της κινητικότητας στα πλαίσια της χορήγησης θεωρήσεων λειτουργούν ευνοϊκά για το σύνολο της αντιπροσώπευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές. Αυτή τη στιγμή υιοθετήθηκε η έκθεση αυτή, περαιτέρω α, ε, επαφές έχουν ε, επαναληφθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει το δικό της βάρος και έχει προβλέψει επίσης περισσότερες θέσεις έτσι ώστε οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λάβουν υπόψη, υπόψη τους τα εξωτερικά τμήματα της εξωτερικής πολιτικής. Αυτοί λοιπόν που ασχολούνται με τα θέματα αυτά θα ασχοληθούν και με τα θέματα της χορήγησης θεωρήσεων. Τώρα θα έπρεπε να τονίσω επίσης ότι αυτά τα απευθύνουμε στα κράτη-μέλη σε δύο επίπεδα στις πρωτεύουσε, γιατί πρέπει και εκεί να διασφαλιστεί ότι τα θα συνδυαστούν τα προξενία και αυτά που κάνουν σε διάφορες υπηρεσίες στα πλαίσια του Σέγγεν. Μπορεί να το θεωρείτε προφανές, αλλά στην πράξη καμιά φορά οι πρόξενοι έχουν ατομικές ιδέες και θεωρούνται ως αφεντικά και ντερβεναγάδες στη χώρα που εργάζονται, χωρίς να σέβονται τους κανόνες εναρμόνισης του Σένιγκεν. Και δεύτερο επίπεδο, τα προξενία που πρέπει να έχουν καλώς εκπαιδευμένο προσωπικό, εκπαιδευμένο μάλλον με συγχωρείτε. και να γνωρίζουν τους κανόνες της συνεργασίας. Τέλος, δεν αφορά τους ανθρώπινους πόρους αυτό το σημείο, αλλά τη συνεργασία μεταξύ ΕΑΣ και Κομισιόν. Οι υπηρεσίες της Κομισιόν που αφορούν τις θεωρήσεις πρέπει να χορηγούν πληροφορίες στο προσωπικό του ΕΑΣ που θα διοριστούν σε διάφορες θέσεις και να γνωρίζουν και αυτοί τα καθήκοντα που έχουν για την τοπική συνεργασία Σέγγιν. Όλα αυτά δεν αφορούν αυστηρά το θέμα αλλά των θεωρήσεων, αλλά θεωρήσαμε στοιχειώδες να κάνουμε αυτές τις συστάσεις και προτέσεις και δεν έχουμε ακούσει και καμία επίκριση από το Συνειβούλιο. Θα θέλαμε βέβαια να ακούσουμε τις απόψεις και της Επιτροπής ΕΛΕΦ για την τοπική συνεργασία ΣΕΝΚΕΝ. Αν θεωρούν ότι μπορεί να γίνουν και άλλες βελτιώσεις, να το ακούσουμε με τα χαρά σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Μήπως η Προεδρία θα ήθελε να προσθέσει τίποτα ή να σχολιάσει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι συντομότατος. Όπως είπε και η Επιτροπή, τα έχουμε αυτά τα δύο θέματα στο πρόγραμμά μας στις 25 Ιανουαρίου. είχαμε. Και έγινε μία ανταλλαγή απόψεων από όλα τα κράτη-μέλη. Δεν καταλήξαμε όμως σε κανένα συμπέρασμα από τις συζητήσεις αυτές. Σκοπεύουμε όμως να το ξαναδούμε. δεν πρόκειται με μία ή δύο συνεδριάσεις να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά θα διασφαλίσουμε ότι η συζήτηση θα γίνει όπως πρέπει. Θα το κρατήσουμε στην ημερήσια μας διάταξη. Κύριε Μάρ, σας κατευχαριστώ για την βαθιά αυτή πληροφόρηση που μας δώσατε. Υπάρχει ένα μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης που είναι που ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση εγώ δηλαδή και θα ήθελα να ρωτήσω πού βασίζεται η ιδέα της συσχέτισης της πολιτικής των θεωρήσεων με την δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά στην καθημερινή ζωή. Μήπως σημαίνει ότι μερικές κατηγορίες θα έχουν προνόμια για τις θεωρήσεις, τι, τι, τι βασίζεται. Και μια, ένα ακόμη σχόλιο. Η προξενική προστασία για την προξενική προστασία χάρηκα που άκουσα ότι θα συμμερίζονται τα βάρη όλοι με το ΕΑΣ για προξενικά θέματα κλπ. Ευχαριστώ. Μόλτερ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γενικό ερώτημα. Η Επιτροπή μας θα συγγράψει έκθεση με συστάσεις προς την Κομισιόν ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα, δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε. Δεύτερο. Είναι επίκαιρο το θέμα και ερωτώ την Κομισιόν. Αν μια χώρα μέλος στο Σέγγεν χορηγήσει βίζα που ισχύει για τις 26 χώρες του Σέγγεν. στείλει μία αντιπροσωπεία της Ένωσης θα μπορέσει να θεωρηθεί ότι οι θεωρήσεις μπορούν να, θεωρούνται και πιο, να γίνονται και πιο κεντρικά αντί από κάθε χώρα μέλος. Ευχαριστούμε κύριε Μόλντορ. Μου λένε ότι το θέμα θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών, η κυρία Στανόκα. Α, ναι, βέβαια, βέβαια. Εμείς στην ομάδα μας πρέπει να συζητήσουμε τη θέση μας για όλα αυτά. Για την κατανομή των καθηκόντων μεταξύ άς και Κομισιόν και φυσικά θέλουμε να υπάρξει μια συνεπής θέση των ομάδων, αλλά αυτά που είπε ο κύριος Μόλτερ ότι πρέπει να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση κεντρικής χορήγησης θεωρήσεων δεν με βρίσκουν συμφώνη. Εμείς θεωρούμε ότι η Κομισιόν δεν είναι και πολύ δραστήρια ή μάλλον οι αρχικές της προτάσεις καλές είναι και φιλοευρωπαϊκές αλλά, αλλά να. Αλλά να, κατά την περαιτέρω εξέλιξή τους, να τώρα στην αξιολόγηση του Σέγγεν και λοιπά, η αμοιβαιότητα της προτάσεις του Κοινοβουλίου, στους φραγμούς που θέτει το Συμβούλιο, βλέπουμε ότι η Κομισιόν δεν επιμένει αρκετά για να αξιολογήσει, για να αξιοποιήσει τις προτάσεις που κάνει με μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ερωτώ λοιπόν, πού, ποιοι είναι οι φραγμοί, γιατί δεν μπορείτε να πετύχετε τις προτάσεις σας. Η Κομισιόν, ο κύριος Ντεκόιστερ. Well, thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, η πολιτική των θεωρήσεων και ο οικονομικός αντίκτυπος την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δείτε ότι εξετάσαμε έγγραφα των G20 και των Υπουργών Εξωτερικών των G20. Υπάρχουν μελέτες οι οποίες δίνουν εκτιμήσεις για τον τουρισμό, για τον ξενοδοχειακό τομέα, για τον τομέα των ε, ταξιδιών. Αν δείτε τα νούμερα αυτά, και δεν λέω ότι τα δεχόμαστε απόλυτα, θα δείτε ότι καθίσταται σαφές ότι εάν αυξηθεί ο ρυθμός των τουριστών, αυτό θα έχει οικονομικά ωφέλη. Και σίγουρα στο μέλλον θα προτείνουμε τροπολογίες και τροποποιήσεις ε, μάλλον στην πολιτική για τις θεωρήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον οικονομικό αντίκτυπο όσων προτείναμε. Φυσικά πρέπει να διεξάγουμε και τη δική μας αξιολόγηση αντικτύπου, όχι βασισμένη σε αυτά που μας έδωσε η συνάντηση των G20, αλλά τα δικά μας. Συνοψίζοντα λοιπόν, χρειαζόμαστε αξιολόγηση αντικτύπου, την οποία φυσικά θα μοιραστούμε με τους συνομοθέτε μας, έτσι ώστε να εξηγήσουμε και να δικαιολογήσουμε τις αποφάσεις που λάβαμε και τη χρονική στιγμή την οποία τις λάβαμε. Και αυτό θα το συνδέσω με την τελευταία ερώτηση Στο στάδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια ανακοίνωση πολιτικής, διότι πιστεύουμε ότι πρώτα είναι καλό να συζητήσουμε με το συνομοθέτη την γραμμή μας για το μέλλον και όταν συμφωνήσουμε με τα διαφορετικά θεσμικά όργανα, τότε αυτό θα μεταφερθεί και θα μεταφραστεί σε συμπαγείς προτάσεις και σε νομικές διατάξεις. Νομίζω όμως ότι είναι επαρκής η πολιτική συζήτηση πρώτα επ' αυτού και μετά να γίνουν πράξεις παρά να αρχίσουμε πρώτα να κάνουμε αλλαγές. Ας συζητήσουμε πρώτα τη γραμμή μας για το μέλλον και μετά ας προβούμε σε πράξεις και αλλαγές. Τώρα, επιστρέφοντας στο συνάδελφο που παρνεύει πρώτος, Αναφερθήκατε στη μία, στην άλλη κατηγορία και το γιατί. Γιατί αυτό που θέλουμε είναι η απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων για όλους τους ταξιδιώτες. Θέλουμε όμως επίσης να κρατήσουμε στοιχεία στην ε, πολιτική αυτή που θα μας επιτρέψουν να ξεχωρίζουμε αυτούς που έχουν καλές και από αυτούς που έχουν κακές προθέσεις και τους να τους κρατήσουμε εκτός. Θέλουμε να υιοθετήσουμε μια συνολική προσέγγιση και όχι να διευκολύνουμε τη διαδικασία ή να την απλουστεύσουμε για μία για την άλλη συγκεκριμένη κατηγορία με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Δηλαδή μας λέμε τώρα ότι θέλουμε να απλουστεύσουμε τη διαδικασία για την Ουκρανία αλλά υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές για, ποιους, για ποιες κατηγορίες ταξιδιωτών, για τους επιχειρηματίες για παράδειγμα που κάνουν επαγγελματικά ταξίδια, για τους τουρίστες θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό επίσης. Δεν είναι το σκεπτικό μας να δώσουμε προνόμια σε λίγους, αλλά σε όλους τους καλοπροαίρετους ταξιδιώτες. Γι' αυτό και υπάρχει το σκεπτικό δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αρχής έκδοσης θεωρήσεων. Εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σήμερα. Όταν αρχίσαμε στο Σέγγεν με την κοινή πολιτική έκδοση θεωρήσεων, ο καθένας είχε τις δικές του προξενικές αρχές Και με το Σέγγεν η θεώρηση αναγνωριζόταν από όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη που είχαν υπογράψει τη συμφωνία. Θα μπορούσε αυτό να μας οδηγήσει σε μια ευρωπαϊκή κοινή αρχή εκδόσεως θεωρήσεων και τον επόμενο χρόνο στην Στοκχόλμη θα το συζητήσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε καθοδόν από τις εθνικές αρχές έκδοσης σε μια κοινή ευρωπαϊκή έκδοση που δεν θα εκδίδει θεωρήσεις εθνικές αλλά ευρωπαϊκές. Έχουμε επίσης και το πλαίσιο κοινή εφαρμογής, το οποίο είναι ένα πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα της έκδοσης θεωρήσεων και αυτό θα μας επιτρέψει να κάνουμε τι. Να έρχονται οι πολίτες, να ζητούν έκδοση θεώρησης και να υπάρχουν τότε αντιπρόσωποι υπάλληλοι των ε, κρατών μελών, κάθε κράτος μέλους, με αρμοδιότητες για τις συγκεκριμένες χώρες. Θα υπάρχει δηλαδή αυτή η γενική αρχή, αλλά θα υπάρχουν και τα επιμέρους ε, στοιχεία της, τα οποία θα είναι αρμόδια για το κάθε κράτος μέλος. Βέβαια αυτό είναι λίγο δύσκολο να γίνει στην πράξη, γι' αυτό και οι αιτήσει σε αυτά τα κοινά κέντρα δεν θα είναι πάρα πολλέ. Γι' αυτό η πρότασή μας για τροποποίηση του κώδικα για τις θεωρήσεις έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα νομικό πλαίσιο έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία περισσότερα από αυτά τα κέντρα κοινή διαχείρισης. Δηλαδή να υπάρχουν αυτά τα κέντρα κοινή διαχείρισης με μία ευρωπαϊκή αρχή που θα τα εποπτεύει. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Έχουμε λοιπόν φτάσει στο τέλος. Επόμενη συνεδρίαση στις 20 και 21 Φεβρουαρίου, όλη τη μέρα και τις δύο ημέρες, Καλό ταξίδι, καλή επιστροφή εύχομαι σε όλους και καλό μεσημέρι.